Κομμάτων της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, άρθρο 135 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Θα ξεκινήσουμε. με το πρώτο σημείο που αφορά την Καμπότζη, τα σχέδια νόμου περί ΚΑΠΑΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Να δώσω τώρα το λόγο στους συντάκτες του εγγράφου αυτού Ο κύριος Έρνεστ Μαραγκάλ, έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε, υποστηρίζουμε αυτό το ψήφισμα και οι υπόλοιποι συντάκτες και ελπίζω και όλες οι πολιτικές ομάδες να συμφωνούν μαζί μας, ανησυχούμε κάπως, έχουμε θορυβηθεί. Διότι περί τίνος πρόκειται, βέβαια είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά γιατί τα βλέπουμε ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνουμε την ε, ανησυχία μας και καταγγέλουμε κάποιες πραγματικότητες, κάποια γεγονότα που... Ε, έχουμε ήδη εξετάσει και έχουμε ασχοληθεί στο Κοινοβούλιο. Πριν από 1,5 χρόνο και λιγότερο ε, είχαμε ασχοληθεί ξανά με την Καμπότζη τον Γενάρη του 2014. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ανεπίλητη αντίφαση και μας ανησυχεί ανάμεσα ε, στην οικονομία, την ευημερία και από τη μια και από την άλλη το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, κάποια στοιχειώδη πρότυπα για κοινωνική νομοθεσία, εργατική κτλ. Τι συμβαίνει τώρα στην Καμπότζη. Υπάρχει μια τριπλή νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που δεν σέβεται καθόλου από ό,τι φαίνεται ούτε τις στοιχειώδεις και ελάχιστες ε, αρχές μας για τη συμμετοχή, για την κοινωνική ε, συζήτηση, τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις αφορά μη κυβερνητικέ οργανώσεις, συνδικάτα κτλ που κανονικά οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να ήταν πρωταγωνιστές των θεμελιδών δικαιωμάτων. Και αυτά όλα συμβαίνουν, ενώ στη χώρα επαναλαμβάνονται ζητήματα που έχουμε δει χαρακτηριστικά τα τελευταία χρόνια, διαφόρων πολιτικών που έχουν να κάνουν με μεγάλες απαλωτριώσεις και εξώσεις μικρών αγροτών ε, από ΓΕΕΣ ε, τις οποίες παίρνει το κράτος για να δώσει παραχωρήσεις και τύπου προβιομηχανικού ας πούμε ε, ή κλείνουν μικρά εργαστήρια, μικρούς τεχνίτες και τα λοιπά. Ένα τμήμα όλων αυτών έχει να κάνει με τις δικές μας απαιτήσεις και κίνητρα που τους δίνουμε. Γιατί ε, ε, ε, υπάρχουν μεγάλες καλλιέργειες και εκμεταλλεύσεις σαχαροκαλάμων που τροφοδοτούν δικά μας αναψυκτικά ας πούμε ή κάποια εργαστήρια βιοτεχνίες που ράβουν ρούχα τα οποία καταλήγουν στα δικά μας μαγαζιά. Λοιπόν, κάνουμε συμφωνίε αλλά τίποτα χωρί δικαιώματα. Nothing without rights. Και όχι να ασχολούμαστε με διάφορα αρχικά και συντμήσει στην νομοθεσία μα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράου. Ένα λεπτό. Grazie, grazie, Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ φανταζόμαι ότι η προπόθεση από την οποία ξεκινάμε όταν συζητάμε για την Καμπότζη είναι ότι εμεί είμαστε ο βασικό χρηματοδότη όλων των αναπτυξιακών έργων που τρέχουν στην Καμπότζη και συχνά έχουμε χρησιμοποιήσει τις ε, ΜΚΑΟ στην Καμπότζη για να εφαρμόσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες ε, ανάπτυξης. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σημαντικό γιατί αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος ο οποίος θα περιορίσει πολύ σημαντικά τις ε, συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις ελευθερίες του συνεταιρίζεστε και το μέσο ουσιαστικά που χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη στην Καμπότζη θα υπονομευτεί. Το ψήφισμα αυτό λοιπόν έχει αυτό το στόχο να μην εγκριθεί αυτή η νομοθεσία γιατί θα στείλει τη χώρα 100 χρόνια πίσω και να γίνει μια προσπάθεια να συνεχιστεί ο διάλογος ε, και να διατηρηθούν τα αναπτυξιακά έργα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Καμπότζη σε ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοράο. Ο επόμενος ε, συντάκτης, ε, ε, ο κύριος Ντεμεσμάκερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Καμπότζη το κυβερνητικό κόμμα θέλει να περάσει ένα νόμο επίμαχο για να φημώσει ε, τα συνδικάτα. Από το 1979 το κόμμα, το λαϊκό της Καμπότζης κυβερνάει και θέλει τώρα να ελέγξει και τις ε, δραστηριότητες και τα οικονομικά των συνδικάτων και το ΜΚΟ γιατί τους θεωρούν αχυρανθρώπους της Δύσης ή του εξωτερικού για να σταθεροποιήσουν την κυβέρνηση ε, ξέρουν ότι χρειάζεται νομοθεσία η ΜΚΟ που είναι 5.000 ε, αλλά δεν θέλουν αυτό το νόμο ο οποίος εγκρυπτό και παραβίστο προετοιμάστηκε ως νομοσχέδιο χωρίς διαβούλευση και πέρασε περίπου νύχτα από το Κοινοβούλιο. Προχτές ακόμα εκατοντάδες ε, ε, άνθρωποι ανήσυχοι διαδήλωσαν γιατί δεν θέλουν να καταργηθούν οι κατακτήσεις τους. Καλούμε την κυβέρνηση να κάνει διαβούλευση, αναθεωρήσει με την κοινωνία των πολιτών ε, την νομοθεσία αυτή και ελπίζω και εμείς να μπορέσουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας με το ψήφισμά μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γερούν Λέναρς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Yes, thank you very much, uh, Chairman, and also thanks to... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Μάλστρομ που μένει μαζί μας ε, το απόγευμα. Είναι πολύ ωραίο που είναι ισχυρή και ενωμένη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια ισχυρή θέση που λέει κατ' ουσίαν ότι εκεί που ανθίζει η κοινωνία των πολιτών, ανθίζει και η δημοκρατία και εκεί που μπορούν να, να λειτουργούν σωστά τα συνδικάτα, ανθίζει η δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ βασικά μηνύματα προ την κυβέρνηση τη Καμπότζη. Πρώτον, αποσύρεται το λόγο για το συνεταιρίζεστε και για τι ΜΚΟ και αποσύρεται το νομοσχέδιο για τα συνδικάτα. Και οποιοδήποτε σχέδιο νόμου στο μέλλον για τους τομείς αυτούς θα πρέπει να αναγνωρίζει τις διεθνώς αναγνωρισμένες ελευθερίες και θα πρέπει να γίνεται δεκτό με μια διαδικασία στην οποία θα συμπεριλαμβάνουν όλοι. Δηλαδή θα γίνεται διάλογος και με τους εμπλεκομένους φορείς στην κοινωνία των πολιτών ε, της μη κυβερνητικής οργανώση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παλώμα Λόπεθ Μπερμέχο για ένα λεπτό έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που απαιτεί να υπογράψει η Κομισιόν επιθετικές εμπορικές συμβάσεις με αναπτυσσόμενες χώρες ε, που διευκολύνει τη δίσδυση των μεγάλων πολυεθνικών στις οικονομίες αυτών των χωρών προσποιείται ότι εκπλήσεται με τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά, δηλαδή την έξωση των αγροτών από τις ε, γέες τους και την εκμετάλλευση των εργατών ε, στα εργοστάσια που εξάγουν τα προϊόντα τους. Απευθύνουμε έκκληση στην κυβέρνηση κυβέρνηση της Καμπότζη να σέβεται τις ε, συμβάσεις ε, του ILO για τα εργασιακά συνδικαλιστικά δικαιώματα που θα επιτρέψει στους εργάτες ε, να αγωνιστούν κατά των πολυεθνικών, να πάψει η απαλωτρίωση από τους μεγάλους ομίλους, τους γεργοδετρέους γεωργοδιατροφικούς. Όμως δεν αρκεί η Ευρώπη να θυμίζει αυτές τις βασικές αρχές. Έχει περισσότερες ευθύνε. για την πλήρη αναγνώριση των ρωσιακών δικαιωμάτων, ε, το δικαίωμα στις γης. Όλα αυτά για να ισχύσουν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στι συμβάσει που υπογράφει με τρίτες χώρες, σε τι αναπτυσσόμενες, γιατί μόνο έτσι θα ανακόψουμε την ε, εκμετάλλευση των εργατών που προς το παρόν απλά και μόνο καταγγέλνουμε. Με τα λόγια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μαριέτε Σάκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, συναδελφοί. Όλοι ανησυχούμε ότι ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών με τις 5.000 συγκεγραμμένες με καπάω στην Καμπότζη μπορεί να υπονομευτεί από την προτινόμενη νομοθεσία που είναι περιοριστική και έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο με το Σύνταγμα αλλά και με τις διεθνείς ε, ε, νομικές δεσμεύσεις ε, που έχει αναλάβει η κυβέρνηση της Καμπότζης με τη δεσμεύσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δαπάνησε 310 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του, θα δαπανήσει μεταξύ του 2014 και 2020. Καλούμε τις αρχές όχι απλά να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και να εκτιμήσουν το ζωτικό ρόλο που παίζουν οι ελευθερίες σε μια ανθούσα ε, κοινωνία των πολιτών ως αναπόσπαστο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, αυτά τα δύο πράγματα πηγαίνουν μαζί και παροτρύνουμε την κυβέρνηση της Καμπότζης να δράσει ανάλογα και να ε, σεβαστεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βάιντεν Χιόλτσαρ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Καμπότζη είναι από τις πιο δοκιμασμένες χώρες του κόσμου Μέχρι 3 εκατομμύρια νεκρούς ε, ε, είχε στα χέρια του το καθεστώς ε, του Πολ Πότ ως εγκληματίες και αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν περάσει και δεν υπάρχει ούτε ευημερία ούτε ελευθερία. Μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισαν να οργανώνονται όλο και περισσότερο οι πολίτες. Ε, το καθεστώς ε, το σημερινό λοιπόν ε, δυστυχώς ακριβώς αυτή τη στιγμή προσπαθεί να περιορίσει και να κλείσει το χώρο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το έχουμε δει και αλλού αυτό σε αναδυόμενες οικονομίες. Αλλά ειδικά για την Καμπότζη και λόγω και της ιστορίας της θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ο εκδημοκρατισμός της χώρας να μην σταματήσει και να μην ε, στραγγαλιστεί από τα σπάργανα. Dank. Ευχαριστώ πολύ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Ταραμπελά. Monsieur député Marc Tarabella, une minute s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδέλφοι έγινε μια προσπάθεια μιας πορείας ε, στους δρόμους της Πομπέγκα ε, για, κατά αυτού του νομοσχεδίου που προβλέπει το, η κυβέρνηση της Γκαμπότζης. Είμαστε με το μέρος τους και θέλω να αναφέρω το θυμό μου για αυτό το νομοσχέδιο που ε, υπορμεύει την ελευθερία έκφρασης πριν από μερικά χρόνια. Κάναμε μια αποστολή ε, στην Καμπότζη με το Κοινοβούλιο για να δούμε ποια ήταν η πρόοδο με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είμαστε οι πρώτοι χορηγοί, οι πρώτοι χρηματοδότε. Ενδιαφέρει την Καμπότζη να έχει αυτή τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναπτυξιακή πολιτική. Πιστεύω ότι πρέπει να οργανώσουμε άλλη μια αποστολή για να μπορέσουμε να ελέγξουμε κατά πόσο συνεχίζουν στη σωστή οδό ή όχι και να τους καταστήσουμε σαφές ότι τους, δίνουμε, τους προσφέρουμε βοήθεια και να πάμε εκεί ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, περνάμε στην διαδικασία Catch Να σας ενημερώσω ότι θα δώσω το λόγο, θα δίνω το λόγο ε, σε ένα άτομο από κάθε πολιτική ομάδα. Ο κύριος Προσπίσμος. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τη συζήτηση αυτή. Παλιά ήμουν και υπεύθυνο για τον νόμο περί δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθε στη χώρα μου είναι δημοκρατικό δικαίωμα για όλους τους πολίτες και πρέπει να επιμείνουμε και η Καμπότζη να εφαρμόσει νομοθεσία που θα συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ώστε οποιαδήποτε ένωση ή ΜΚΟ, αν πληρεί τις νομικές προϋποθέσεις, να μπορεί να καταχωρίζεται και να μπορεί να ιδρυθεί χωρίς το κράτος να μπορεί να το αποτρέψει αυτό στην Καμπότζη. Είναι πολύ καλό να το πούμε και να το συσχετίσουμε και με τη χρηματοοικονομική βοήθεια που στέλνουμε στην Καμπότζη. Μόνο αν αλλάξει την νομοθεσία της η Καμπότζη θα πρέπει να μπορεί να έχει δικαίωμα και για τη συνέχιση της, της ε, χρηματοοικονομικής βοήθειας. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ο κύριος Φρουντζούλικα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για τα νομοσχέδια ε, της κυβέρνησης της Καμπότζης με τα οποία περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης του συνεταιρίζεστε, του συνέρχεστε θα παραβιαστεί δε και το Σύνταγμα. Ε, με τον τρόπο αυτό θα συρρυκνωθεί ο χώρος που, ε, που υπάρχει για την κοινωνία των πολιτών. Αυτό το σχέδιο για τις ενώσεις και τις ΜΚΟ θα πλήξει σοβαρά τις ΜΚΟ που εργάζονται επί τόπου και την ε, συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ της Καμπότης αλλά και τα αναπτυξιακά προγράμματα της Ένωσης και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα τελευταία 30 χρόνια την Καμπότζη για την ανοικοδόμηση ανασυγκρότηση. Είμαστε ο σημαντικότερο εταίρος ε, παροχής ε, αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεμελιωδών ελευθεριών και με βάση και την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα πρέπει η κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ Ιβάν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από τα όσα έχει περάσει η Καμπότζη, τους πολέμους και τις τραγωδίες, περιμέναμε η χώρα αυτή να σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά φαίνεται να πηγαίνει προς τα πίσω αντί για προς τα μπρος η απαλωτρίωση γεών, η αρπαγή γεών, ε, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα όσα γίνονται κατά τον ΜΚΑΠΑ, ο, ο και κατά της ελευθερίας ε, του συνεταιρίζεσθε και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, από ό,τι φαίνεται η Καμπότζη πήγαινε προς τα πίσω. Εμείς ε, εκφράζουμε την συμπαράστασή μας σε αυτή τη χώρα και ελπίζουμε να συνεχίσει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει να θέσει ισχυρές αρχές. Έχουμε το δικαίωμα και πρέπει να τους απαιτήσουμε από αυτούς να συμπεριλάβουν στην νομοθεσία τους τα θεμελιώδη δικαιώματα στα οποία εμείς πιστεύουμε. και τη διατήρηση των βασικών ελευθεριών στις οποίες ε, περιμένουμε. Ο κύριος Φάβιο Μασίμο Καστάλτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία τριπλή προσπάθεια προσβολής ε, της ε, ελευθερίας των βασικών δικαιωμάτων, ε, προσβολής των διεθνών οργανισμών και των δικαιωμάτων των συνδικάτων. Ο Πρωθυπουργός της Καμπότζης κινείται προς ένα αυταρχικό καθεστώς και ένδειξε αυτό αποτελεί αυτή αυτή η νομοθεσία όπως και η νομοθεσία που θα κάνουν για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που ακόμη δεν γνωρίζουμε αλλά που επίσης θα πλήξει την ελευθερία του λόγου online. Εμείς ως βασική χορηγοί θα πρέπει να πετύσουμε πολλά από την Καμπότζα αλλά και από εμάς τους ίδιους ώστε να διασφαλιστεί η δική μας εμπορική πολιτική σε συνοχή με τη συμπεριφορά των δικών μας πολυεθνικών που να μην πηγαίνουν και να εφαρπάζουν τις γέες των Καμποτζιανών με τέτοιες κινήσεις αυταρχικές. Το σύμφωνο ε, ελεύθερων, ε, ελευθεριών και πολιτικών δικαιωμάτων μας υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα του συνεταιρίζεστε και οι ελευθερίες δεν είναι διαπραγματεύσιμα αλλά θέλουμε δράση από την Κομισιόν που να απαιτήσει από την κυβέρνηση της Καμπότζη να επαναχωρήσει αμέσω από αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κριστίνα Μόρβα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα να προκαλέσω κάποιον, αλλά ε, με αγάπη αντίθετα ε, μιλώ όπως μιλώ. Και ελπίζω να έχει και τα ακουστικά της η Επιτρόπος, γιατί στρέφομαι στην ίδια να τη ρωτήσω. Αν με ακούει. Α, με ακούει, ωραία. Κυρία Επίτροπε, έχετε ακούσει την επόθεση «Γιούντιτ Σίμα είναι ηγέτης, ε, ή υπήρξε ηγέτης ε, ε, συνδικαλιστικού κινήματος στην Ουγγαρία, πάρα πολύ δημοφιλής και μόλις καταδικάστηκε σε τριετή κάθυρξη λόγω των δραστηριοτήτων της ως ε, του συνδικαλιστικού κινήματος. Ήταν στην αστυνομία, ήταν δικαλίστρια ε, και έγινε πάρα πολύ γνωστή όταν είχαν γίνει πριν από κάποια χρόνια πολύ βίες συγκρούσεις ε, της αστυνομίας με διαδηλωτές. Είχε ζητήσει να μην ε, ακολουθήσουν ε, οι αστυνομικοί συναδελφοί της τις εντολές ε, και είναι γελίο να μπορεί να διώκεται ένας άνθρωπος σήμερα για αυτό το λόγο σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάλστρομ τώρα, η Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, συζητούσαμε την Καμπότζη από την Ουγγαρία να τη συζητήσουμε μια άλλη φορά. Όπως πολύ επισημάνατε, η Καμπότζη έχει πραγματικά μια πολύ δραστήρια κοινωνία των πολιτών και πολλέ ε, ΜΚΟ και ε, οργανισμοί δραστηριοποιούνται σε πολλού τομεί και η κυβέρνηση, όπω γνωρίζετε, εδώ και πολλά χρόνια λέει ότι χρειάζεται μια νομοθεσία για το συνεταιρίζεστε ώστε να υπάρχει διαφανή νομοθεσία για τον τομέα. Εμεί παρακολουθούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όλο το θέμα πολύ στενά. Από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η ιδέα για την νομοθεσία αυτή πριν από πολλά χρόνια, τα νομοσχέδια ε, ε, έχουν συζητηθεί σε άτυπε και επίσημε συναντήσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καμποτζιανή κυβέρνηση. Η αντιπροσωπεία μα και ο πρέσβη μα ε, έχουν τακτικέ επαφέ σε διάφορα επίπεδα ώστε να εκφράζουν τι σαφεί απόψει μα και να έχουν γίνει κατανοητέ από την κυβέρνηση. Και του καταστήσαμε σαφέ ότι μια τέτοια νομοθεσία θα πρέπει να επιτρέπει και όχι να περιορίζει την ελευθερία του συνεταιριστή και τη έκφραση στην Καμπότζη. Επισημαίνουμε ότι μια δημοκρατική διαδικασία πρέπει να είναι διαφανή και να συμπεριλαμβάνει πλήρη διαβούλευση με όλου του ενδιαφερομένου. Η νοοτροπία διαλόγου αποτελεί βάση για κάθε δημοκρατία. Με την αντιπολίτευση, την κοινωνία των πολιτών, με τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο μέσω ενό τέτοιου διαλόγου μπορεί η κυβέρνηση να λάβει υπόψη τι ανάγκε και τι ανησυχίε των όσον αφορά η νομοθεσία. Μια διαδικασία χωρί αποκλεισμού επιτρέπει σε μια κυβέρνηση να ψηφίζει νόμους που πραγματικά είναι προς το συμφέρον των ανθρώπων. Η Εθνοσυνέλευση τη Καμπότζη έχει να παίξει σημαντικό ρόλο εδώ. Οπότε καλωσορίζουμε την απόφαση τη Εθνοσυνέλευσης να διοργανώσει διαβουλεύσεις επί του νομοσχεδίου για τις ΜΚΠΑΟ. Και ορισμένε διαβουλεύσει έχουν ήδη ξεκινήσει και ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά του ε, θα αποτυπωθούν στο κείμενο του νομοσχεδίου. Φυσικά είναι σημαντικό να υπάρξουν ε, συναντήσει μεταξύ ομοτιμών, μεταξύ μελών του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Εθνοσυνέλευση τη Καμπότζη, ώστε να του βοηθήσουμε να ενισχύσουν τη δυνατότητά του, να εξετάζουν ε, διεξοδικά και να βελτιώνουν την νομοθεσία σε στενή επαφή με την κοινωνία των πολιτών και με ένα πνεύμα διαλόγου. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και τι εξελίξει, διότι σε εποχέ όπου η κοινωνία των πολιτών και τα συνδικάτα αντιμετωπίζουν ε, πολλές πιέσεις, περιορισμούς και εμπόδια σε πολλές χώρες. Η Καμποτζή έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι πραγματικά έχει δεσμευτεί να ενισχύσει ε, τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. Έχω λάβει 7 προτάσεις ψηφίσματος από τους πρασίνους, η FDD, η ECR, ΕΛΚ, Σοσιαλιστών Δημοκρατών, ΓΟΕ.